Έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος της Επιτροπής ΔΕΒΕ, το οποίο θα ψηφιστεί αύριο. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει αύριο, ημέρα 5η, 26 Νοεμβρίου. Θα ξεκινήσουμε στις 9 η ώρα. Έχει την ημερήσια διάταξη στο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λίγη εδώ η συνεδρίαση. Καλό βράδυ.